Θα ξεκινήσω, συνάδελφοι. Να κάνω μια ανακοίνωση πρώτα. Να σας πληροφορήσω ότι τη Δευτέρα μαζί με τους Πρόεδρους του Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 40 74 ο Πρόεδρος θα υπογράψει έξι νέες νομοθετικές πράξεις. Οι τίτλοι των πράξεων αυτών θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά της παρούσης συνεδριάσεως. Θα ήθελα όμως να καθίσετε, να μην καθυστερήσουμε άλλο, τις ψηφοφορίες που έχουμε. Να διευκρινίσω επίσης ότι δεν θα διαβάζω τους αριθμούς, δεν θα σας μεταφέρω τα αριθμητικά αποτελέσματα, δεν θα σας λέω ούτε καν ευχαριστώ. Το πρώτο θέμα είναι η ψηφοφορία μέσω της απλοποιημένης διαδικασίας του άρθρου 138 του κανονισμού για την έκθεση του κυρίου Σκέρια για το έτος του εθελοντισμού. Ο εισηγητής θα ήθελε το λόγο. Ο κύριος Κούρια. Πάρα πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Να ευχαριστήσω όλους του συναδέλφους για τις προσπάθειές τους, να ευχαριστήσω όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές που εργάστηκαν, όλους τους σκιώδεις εισηγητές και τους εισηγητές που έχουν προσφέρει στην έκθεση αυτή. Νομίζω ότι εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο του εθελοντισμού. 100 εκατομμύρια